Οι περιστάσεις είναι ιδιαίτερες γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταρτήσουμε, να εκπονήσουμε τον προπολογισμό αυτό, όχι μόνο όμω με αριθμητικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσω του προπολογισμού να θέσουμε τι πολιτικέ μα προτεραιότητε. Θέλουμε ένα προπολογισμό, ο οποίο θα προβλέπει επενδύσει στα πλαίσια μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού. Αυτό είναι δυνατό και μπορεί να μην αρέσει στους λαϊκιστές, σε όλους αυτούς που προωθούν μια ρητορική γεμάτη ψευδείς ειδήσει και ψευδή στοιχεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά την εισηγήτριά μα, τη Μόνικα Χολμαϊρ, η οποία δεν με ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά θα με ακούσει σε λίγο ελπίζω, διότι στην έκθεσή της κάνει πολύ ποιοτικέ προτάσει, οι δημοσιονομικέ της προτάσεις και προοπτικέ, αγαπητή Μόνικα, επέτρεψαν να καταλήξουμε σε επικοδομητικούς συμβιβασμού. Και θα ήθελα, σε ευχαριστώ Μόνικα, αυτό έλεγα, και ήταν ε, πολύ σημαντικό για όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαμε στην εκπόνηση έκθεσης αυτής να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προπολογισμού αυτού. Εγώ εργάστηκα εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας για τα εξή θέματα, τις εξή προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα να αυξηθεί η κοινωνική διάσταση του προπολογισμού αυτού, να υπάρχει απαραίτητη εποπτεία όσον αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και βοηθά χιλιάδες νέους οι οποίοι βρίσκονται σε άτυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι του προπολογισμού αυτών υπάρχουν τα απαραίτητα κοινωνικά πρότυπα. Επίσης, προωθείται η πολιτική Τη ενσωμάτωση και την κατάργηση τη διακριτική μεταχείρισης. Θέλουμε επίση να προωθήσουμε την πολιτική για του νέου, για τον πολιτισμό, προγράμματα όπω το Εράσμου, το Μίντια ή τη Δημιουργική Ευρώπη. Θέλουμε να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου πολίτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να τηρήσουμε τη δεσμεύση τη ΜΑΠΣ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Και κάτι ακόμα όμως θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ακόμα περισσότερο ενδεχομένω, όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει εδώ πέρα να ασχοληθούμε με τις μεταναστευτικές ροές και με την πολιτική αναπτυξιακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες δηλαδή, αλλά να δούμε τι γίνεται επίσης και στο στερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να προκαλείται σύγχυση με την πολιτική ασφάλεια που είναι εξίσου σημαντική. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό προληπτικά να καταφέρουμε να προβλέψουμε κάποια κονδύλια σε σχέση με όλες τις εξελίξεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι. Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και πρέπει να στραφούμε κατά τη στασιμότητα, όπω είπε πριν από λίγο και ο επίτροπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλισμούς με αλληλεγγύη για όλου. Μια ακόμα προτερότητά μα είναι να αποφύγουμε μια κρίση πληρωμών, αυτό το είπε και ο επίτροπο πριν από λίγο, και δεν σα κρύβω ότι οι τελευταίε πληροφορίε που λάβαμε όσον αφορά το Brexit προφανώς μας δημιουργούν πραγματικές ανησυχίες. Τέταρτη προτεραιότητα είναι η χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων, των ρητρών ευελιξίας, όπως προβλέπεται από τον υφιστάμενο δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να έχουμε ένα πραγματικά ευέλικτο προπολογισμό. Θα πρέπει το Συμβούλιο να λάβει τις ευθύνες του. Το να είναι θεωρητικά και μόνο υπέρ της Ευρώπης είναι πολύ αξιόλογο σίγουρα, αλλά στην πράξη έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε, η πρόταση αυτή για τον προπολογισμό του 2020 που σας παρουσιάζουμε σήμερα δεν είναι μόνο υπεύθυνη, αλλά αποτελεί πραγματική γέφυρα προς το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλοι μας λοιπόν, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως το Συμβούλιο, είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να καταστήσουμε έμπρακτο τον προπολογισμό αυτό. Ευχαριστώ κύριο Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, Συνάδελφοι. Είναι μάλλον τελευταίος μου προϋπολογισμός. Σίγουρα πάντως είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που τα σημερινά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα προετοιμάσουν κατά τη διάρκεια αυτή τη θητείας. Είναι ο τελευταίο επίση προπολογισμό του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο και μαζί με το Brexit ε, θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε. Όμως δεν έχουμε χαλαρώσει, χάρη στην κυρία Χολμάγερ. Την στηρίζουμε σε ό,τι αφορά τον, τον προσανατολισμό και τις προτεραιότητες για, για το 2020. Ανεφόρον, επιθυμούμε να τεθούν στη διάθεσή μας τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να στηριχθούν οι επενδύσει, στρατηγικέ επενδύσει, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα, την τεχνητή νοημοσύνη, υπέρ τη οικονομική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία θέσεων εργασία ποιότητα, ποιοτικών θέσεων εργασία. Στηρίζουμε επίση το αίτημα για περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα, για προγράμματα όπω το COSME, ε, που βοηθούν τις startup και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την ενίσχυση τη χρηματοδότηση του Erasmus Plus, ε, της πρωτοβουλίας για τους ε, νέους και του προγράμματος αλληλεγγύης. 93.000 ήδη αιτήματα, 93.000 αιτήσει από νέους έχουν ήδη παραληφθεί. Συγχαρητήρια. Επίσης, ανάγκη να προβλέψουμε από το 2020 τι ε, τις απαραίτητες πιστώσεις πληρωμών για να αποφύγουμε ε, το, το μεγάλο όγκο πληρωμών που χρειάστηκε να συσσωρευτούν την προηγούμενη περίοδο 2014 και μετά. Δυστυχώ, το Συμβούλιο δεν δείχνει ευαισθησία εναντί των προβλημάτων που αυτές οι καθυστερήσει έχουν δημιουργήσει σε επιχειρήσεις αλλά και στα κέντρα έρευνας. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση για την καλύτερη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, ε, να καταπολεμήσουμε τους λαθρεμπόρους ε, ανθρώπων και να βελτιώσουμε τις υποδομές υποδοχής των ανθρώπων που χρειάζονται την προστασία μας ε, και στους οποίους έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε άσυλο. Χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια επίσης στην ενίσχυση της ασφαλείας μας. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας ασφάλεια, να χρειαζόμαστε ε, να δώσουμε τα κατάλληλα μέτρα μέσα συγγνώμη, στις υπηρεσίες στους οργανισμούς που έχουμε δημιουργήσει με, σεβασμό, με το πλήρη σεβασμό, σεβασμό βέβαια στα, στα δικαιώματα των πολιτών μας. Επίσης, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις ε, προσπάθειες ε, για να συντονίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την άμυνα μας. Τρεις ακόμα ανησυχίες έχω. Η έρευνα και η καινοτομία, όπως όλοι είπατε, είναι η βάση για την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών μας στο μέλλον. Το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε αρκετά. Η σημερινή Ευρώπη έχει ξεπεραστεί από την Νότιο Κορέα, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και πολύ σύντομα και από την Κίνα σε ό,τι αφορά το ποσοστό ΑΕΠ που αφιερώνεται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν κατανοώ και δεν δέχομαι την άποψη ε, του, τη συμπεριφορά του Συμβουλίου που αρνείται την εφαρμογή του άρθρου 15.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις του ε, ορίζοντος Ευρώπη ε, την επόμενη χρονιά εξαιτία του γεγονό ότι ορισμένα προγράμματα δεν χρηματοδοτήθηκαν επάρκώ. Επίσης υπάρχει το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι νέοι έχουν βγει στους δρόμους το προκυρήσουμε, ε, τον αγώνα αυτό παντού, αλλά δεν κάνουμε αρκετά. Κατά τη διάρκεια της περίοδου 2014-2020 δεν αφιερώσαμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση κλιματική κλιματικής το 20% του συνολικού προϋπολογισμού που είχαμε ε, αποφασίσει να αφιερώσουμε. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να αλλάξει. Επίσης, χρειάζεται να στηρίξουμε τον οργανισμό των Εθνών που ε, βοηθάει τους πρόσφυγες στην Παλαιστίνη. Ο Ντόναλτ Τραμπ απέσυρε την βοήθεια των ΗΠΑ, τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ στην UNRA. Ε, δεν πρέπει και εμείς να γίνουμε εξίσου κακοί με τον κύριο Τραμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σολέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση για τον προπολογισμό του 2020 στις Καθηγητήρια γραμμές, δηλαδή είναι ο τελευταίο προπολογισμό του τρέχοντος ΠΔΠ, Ένα προπολογισμό που θα πρέπει να είναι γέφυρα για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο από πολλέ πλευρέ, είναι καλό σημείο αφετηρία για τι ε, επικείμενες διαπραγματεύσει. Για παράδειγμα, η έκθεση σωστά εκφράζει την ε, δυσαρέσκειά του γιατί δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για, τους, για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή και δεν ε, φτάνουμε καν στο 20% που είχαμε πει ότι θα δαπανούμε σε σχέση με το κλίμα. Σήμερα είχαμε εδώ νέου ακτιβιστέ για το κλίμα και συζητήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει δράση κατά τη κλιματική αλλαγή. Αυτοί οι κινητοποιημένοι νέοι μα καλούν να δράσουμε, να έχουμε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη που να βασίζεται στι ανανεώσιμε και αυτό να γίνει τάχιστα. Όμω, δεν προχωράμε. Ούτε αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, ούτε για να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα. Και ο χρόνος μας πιέζει. Γι' αυτό θέλουμε ένα πολύ πιο πράσινο προϋπολογισμό. Πρέπει το κλίμα να είναι στη βάση όλων των πολιτικών μας και να ελέγχονται εάν ε, είναι σύμφωνε με τους στόχους των ε, Παρισίων και με τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Επίσης, σωστά καλή για περισσότερε κοινωνικέ κοινωνικές φιλοδοξίες. Χωρίς κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει ένωση ισοτήμων πολιτών. Χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου για την πρωτοβουλία, για την απασχόληση των νέων, για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, για την ένταξη των μεταναστών. Και περισσότερα πρέπει να κάνουμε για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Γιατί και αυτά είναι ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Θετικό είναι ότι ο... η έκθεση αυτή λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την κοινοτομία, την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική μεταμόρφωση της οικονομίας. Αλλά λέει ότι η άμυνα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτές οι δαπάνες που πολλοί θεωρείται προτεραιότητα δεν θα είναι αποτελεσματικές. Δεν θα, τα, δεν θα αντιμετωπίσουμε έτσι τα θέματα του κατακαιρματισμού και ε, του πλεονάζοντος δυναμικού. Έχουμε πολύ πιο πήγος προτεραιότητες για να καλύψουμε τον προβλησμό της Ένωσης. Τέλος, κάτι διαδικαστικό τα μέλη της Επιτροπής Μπούτς και ο Επίτροπος Ότιγκερ θα θυμούνται τι έγινε με το 15.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού κατά την τελευταία συνδιαλλαγή. Τώρα από την αρχή των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό λέμε σαφέστατα ότι θέλουμε να χρησιμοποιηθεί αυτό το άρθρο. Και δεν θα πρέπει να μας κορυδέψετε για άλλη μια φορά. Κύριε Σολέ, υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Έθεριτζ. Τη δέχεστε? Ναι. Κύριε Έθεριτς. Ευχαριστώ που τη δεχτήκατε. Ε, πραγματικά θέλω να μου πείτε τι θέλετε. Θέλετε για πολλά σημεία περισσότερα. Είναι ένας προϋπολογισμός που συνεχώς αυξάνεται. Πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που ο προπολογισμό θα μπορούσε να μειωθεί, τουλάχιστον να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Ή νομίζετε, όπως ε, στο σκέτ των ε, Monty Python ότι μπορείτε να καταπίνετε όλο και περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων μέχρι που να σκάσετε. Ε, θεωρείτε ότι μπορεί να συνεχίσει να ε, αυξάνεται ο προπολογισμό τη Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Ίσως για τις λεπτομέρειες του επόμενου ΠΔΠ, φυσικά οι προπολογισμοί δεν μπορούν να αυξάνονται συνεχώς γιατί οι πόροι είναι περιορισμένοι. Αλλά ένας προπολογισμό έχει δύο πλευρές. Έσοδα και δαπάνες. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται για τα έσοδα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε σταδιακά, όχι με απότομα άλματα, να αυξήσουμε τους πόρους του προπολογισμού της Ένωσης. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εσείς δεν το πιστεύετε. Και γι' αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου. Μεγαλύτερο προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Η κυρία Νι Ριάντα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα τουλάχιστον να έχει την ευγένεια ο επίτροπο να μ' ακούει. Είναι πολύ σημαντικό αντί να μιλάτε στο τηλέφωνο να ακούτε του ευρωβουλευτέ. Είναι προσλητικό το ότι δεν μα ακούτε και την ε, επόμενη φορά που θα έρθετε στην Επιτροπή μας θα φροντίσουμε και εμείς να μην σας ακούσουμε. Τέλος πάντων. Μόλον ότι αποφασίσετε τελικά να μην ακούσετε, θα απευθυνθώ στους υπόλοιπους συναδέλφους. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την έκθεση αυτή της κυρίας Χολμάιερ για όλη την εργασία που έχει εμπλουτίσει την έκθεση αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που δικέ μου γίνανε δεκτέ, που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση των προγραμμάτων PIS και Interreg και ελπίζω ότι η υποστήριξη αυτή θα συνεχιστεί, γιατί αντιμετωπίζουμε πάρα πολλέ προκλήσεις εξαιτία ε, του Brexit. Πρέπει βέβαια να πω ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα καμία αναφορά επαρκής για την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολλά κονδύλια δίνονται στην άμυνα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να δίνουμε πάρα πολλά κονδύλια στην άμυνα τον θέμα αρχή. Πάντω το ζήτημα αυτό θα το συζητήσουμε περισσότερο και στα πλαίσια τη Επιτροπή. Οι ελίε μα επίση αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ προκλήσει, το ίδιο και οι αγρότε μα και καθότι, όπως είπα πριν από λίγο, υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια έκτα της ανάγκης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Brexit. Στα σχέδια αυτά δεν είδαμε κάτι όμως το τόσο ουσιαστικό, γιατί εντάξει, πολύ ωραία, αναφέρεστε στις αεροπορικές μεταφορές, μπορεί να έχουμε αεροπλάνα, αλλά δεν έχουμε αλεξίπτωτα. Τα πάντα εξαρτώνται ουσιαστικά από την καλή βούληση των Βρετανών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνούν σε πάρα πολλά σημεία, άρα βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Στην πράξη, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε ω Επιτροπή Προπολογισμών πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που προκύπτουν από το Brexit. Φτάνουμε όλο και πιο κοντά στην ημέρα της αποχώρησης. Από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για να χρηματοδοτήσουν τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελείωσε η παρέμβασή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που να με ακούσετε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Δεν με νοιάζει που επίτροπος ε, τηλεφωνάει. Είναι πολύ φιλόδοξος αυτός ο προϋπολογισμός. Πρόσθετη χρηματοδότηση πολλών πραγμάτων. Εράσμος, παίρνει πολλά περισσότερα. Ελεύθερη κυκλοφορία, περισσότερα. Ε, διοικητικός προϋπολογισμός και βέβαια στρατιωτικές δαπάνες. Κάτι μας είπαν ότι είναι φανταστικό και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πραγματικότητα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι μας λέγανε. Στην παράγραφο 28 όμω. υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληρώσει για τη συμμετοχή του σε αυτά τα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή κανένα δεν ξέρει τι θα συμβεί. Ναι, η Τερέσα Μέη πανηγυρίζει παρόλο που δεν ξέρει τι κάνει. Οπότε ίσως πραγματικά κάνετε καλή πρόβλεψη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και το χάος αυτή τη στιγμή. Όποιο ανοίξει το κοινοβουλευτικό κανάλι του BBC ή διαβάσει μια βρετανική εφημερίδα, βλέπει ότι επικρατεί χάος. Και πολύ πιθανό όλα αυτά τα κόμματα με τους αδύναμους ηγέτες να διαλυθούν στα εξών συνετέθησαν. Και μπορεί τελικά κάποιος να βρεθεί που να ακούσει τι λέει ο λαός και, δεν και λέει ότι δεν θέλει να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια λίρες αποχαιρετισμού όταν έχουμε τόσα απλά προβλήματα στη χώρα μου. Καταλαβαίνω γιατί πληρώνεται τόσα πολλά λεφτά περιμένοντας ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει στον προπολογισμό, αλλά νομίζω ότι είναι τυχερό παίγνιο. Ποντάρεται σε κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο. Προσέξτε, γιατί οι Βρετανοί μπορεί να πούνε νό. Συζητάμε εδώ την κατάρτιση του προπολογισμού 2020. Ένας ιδιαίτερα δύσκολος και πολύπλοκος προπολογισμός για το σύνολο της Ένωσης. Μα για ακριβώ αυτό το λόγο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Χολμάιερ η οποία αποφάσισε να αναλάβει αυτό το τόσο δύσκολο έργο. Είναι καταρχάς ο τελευταίος προπολογισμό στο πολιτισμο δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να καταβάλουμε πάρα πολλές πληρωμές σε τιμολόγια που καταρτίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Το 2020 θα έχουμε αυξημένες δαπάνες, αφού το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ένα άλλο λόγο που είναι δύσκολο προπολογισμό αυτό είναι γιατί συνήθω το τελευταίο έτο, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το επιπλέον πρόβλημα του Brexit. Και όπως είπε ο σας, αντιμετωπίσουμε μια χαοτική κατάσταση. Καλούμεθα λοιπόν να εκπονήσουμε έναν προπολογισμό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε απρόβλεπτες, ακόμα και χαοτικές καταστάσεις. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονό ότι ενδεχομένω ο προπολογισμό αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να τροποποιηθεί με βάση την εξέλιξη που θα πάρουν τα πράγματα όσον αφορά το Brexit. Επίση, ο προπολογισμό αυτός εκπονήθηκε παράλληλα με την όλη εργασία που γίνεται για το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και το ενδιαφέρον με τον προπολογισμό αυτό είναι ότι ε, εισάγει ήδη από το 2020 κάποια νέα στοιχεία τα οποία, εμείς, τα οποία θα μας απασχολήσουν για πολλά χρόνια μετά το 2020. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μελλοντικό προπολογισμό, ο οποίο καταρτίζεται ήδη από σήμερα. Πράγματα τα οποία από τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε χωρί να περιμένουμε το 2021 ή τα επόμενα έτη. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική ανάπτυξη, όπω ο Horizon 2020 και το πρόγραμμα Erasmus. Μιλάμε όλο και περισσότερο για την ενίσχυση του προγράμματο αυτού. Λέμε ότι θα πρέπει να τριπλασιαστεί ήδη από το 2021 ο προπολογισμό του. Αυτό όμω ξεκινάει ήδη από το 2020 ω πρόθεση. Ασχολούμεθα επίση ε, και με άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, την ε, ανθεκτικότητα κάποιων ταμείων που έχουν να κάνουν ε, με την άμυνα. Το 2020, αν θέλετε, είναι ένα προπαρασκευαστικό έτος για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι απλώς το τελευταίο έτος μιας δημοσιονομικής περίοδου. Όταν μιλάμε επίσης για καινοτομία, Ήδη από το 2020 υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το Brexit, όπως είπαμε. Αλλά έχουμε αυξημένες δαπάνες και ουσιαστικά το 2020 είναι ο προπολογισμό αυτό ένα προπολογισμό γέφυρα ανάμεσα στα δύο πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια. Ένας προπολογισμό λοιπόν που βρήθη προκλήσεων και που θα καθορίσει πάρα πολύ το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ κυρία Τόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη Μόνικα Χολμάιερ που πραγματικά μας άκουσε και έκανε τους αναγκαίους συμβασμούς. Ο προπολογισμό 2020 είναι το τελευταίο βήμα του πολιτού πλαισίου και για άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο θα δεσμευθεί με αποτελεσματικότητα και πεποίθηση ότι θα επιβάλλει τις προτεραιότητές του. Ε, και αγαπητέ κύριε Έθεριτζ, λυπάμαι. Α, έφυγε. Α, έφυγε κρίμα. Εν πάση περιπτώσει, αντίθετα από αυτά που ισχυρίζεστε, ο προορισμός της Ένωσης ε, μειώνεται από δεκαετία του 90 και μετά. Κύριε Επίτροπε, Απευθύνομαι σε εσά, γιατί πολύ θα ήθελα να ασφάλω, να μπορούσα να πιστεύω να σταματήσει αυτή η παράλογη διελκυστίδα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Θα ήθελα πραγματικά, διακαώς θα επιθυμούσα, η Επιτροπή να μην ε, είναι σε αυτή την διακυβερνητική λογική όσον αφορά τον προπολογισμό. Θα να μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι το Κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει αυτό τον προπολογισμό μόνο εάν αυξηθεί η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της χρηματικής αλλαγής όπως είχαμε αποφασίσει για το πολιτές πλαίσιο 14-20. Πολύ θα ήθελα ο προπολογισμός του 2020 να χρηματοδοτήσει την ένταξη των ε, μεταναστών και των ε, ε, ετούντων άσυλων και να μην χρηματοδοτεί την εξωτερικοποίηση την υπεργολαβία στην πολιτική μας για τους πρόσφυγες. Θα ήθελα να βοηθάει ο προβλημός αυτός το ευρωπαϊκό εγχείρημα και οι νέες προκλήσεις να έχουν νέους πόρους διάθεσή τους. Το Κοινοβούλιο να μην δέχεται οι νέες προτεραιότητες να χρηματοδοτούνται εις βάρος των πολιτικών αλληλεγγύης. Πόσο θα ήθελα το Brexit να μην αξιοποιείται άλλη μια φορά ως πρόσχημα για να μειωθεί ο προβλημός της Ένωσης. Θα ήθελα πολύ να σας πείσω για όλα αυτά ότι δεν δίνουμε αρκετά για την ισότητα των φύλων στον προπολογισμό και ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Καταλήγω λέγοντας ότι εύχομαι στην κυρία Χολμάιερ κουράγιο αν θέλει να υπάρξει ένας προπολογισμό στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Για να μην ε, πάρουμε μόνο ψίχουλα. Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάραντ. Έχω γραμμένα κάποια σημεία για την ομιλία μου που λένε ότι οι σημαντικές προτεραιότητες έχουν περιληφθεί κλιματική αλλαγή, απασχόληση, έρευνα και το κλειδί είναι η άμυνα. Εδώ θα βάλω στην άκρη τη σημειώση μου και θα πω ότι ε, δεν με ανησυχεί τόσο πολύ η δαπάνη για, τις, για την άμυνα γιατί η καλή άμυνα μπορεί να μας χρησιμεύσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους. Και ίσως όχι τόσο πολύ για τον προϋπολογισμό. Αντίθετα με την κυρία Νιριάντα και τον κύριο Έθριτζ που είπαν ότι ο Επίτροπος δεν ακούει. Να πω ότι ο κύριος Έτιγκερ έπαιρνε πληροφορίες για τον Brexit από το αριστερό του αυτή και μας άκουγε εμάς από το δεξί του αυτή. Οπότε, κύριε Έθριτζ, εσείς που είστε αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων να που είστε εδώ, όχι βέβαια. Ε, δεν θα γίνεται. επίτροπο αν δεν μπορείτε να κάνετε multitasking. Τέλο πάντων, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό να πω το εξή. Ήταν μεγάλη τιμή να θητεύσω στην Επιτροπή Προπολογισμού και να μάθω από τον κύριο Ντεπρέ, τον κύριο Ολτμπριχτ, τον κύριο Φερνάντε, από την Μόνικα Χολμάιερ και από την κυρία Γκαρδία Θάβαλ και άλλου. Τελικά βέβαια δεν καταφέραμε όσα περιμέναμε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και τη χρηματοδότησή τους. Την Παρασκευή τα σχολεία απεργούν για την κλιματική αλλαγή στην Εστονία για πρώτη φορά. Ο γιος μου θα συμμετάσχει. Ο πατέρας μου, επίσης παλιό μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, θα είναι εκεί και ως κλιματολόγος. Εγώ που θα πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαι. Ασφαλώς και εγώ θα είμαι μαζί τους. Γι' αυτό το λόγο θα υποστηρίξω την τροπολογία της, των φιλελευθέρων που κάνει μια, ε, συνδέει την Συμφωνία του Παρισιού με τις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες. Μπράβο στους φιλελεύθερους. Τελειώνω. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει κύριε Πρόεδρε. Ο οποίο είπε ο κ. Διπρέ μπορεί να είναι ο τελευταίο του προπολογισμό και εμένα μπορεί να είναι ο τελευταίο μου προπολογισμό. Και είναι τρομακτική, αλλά για την κλιματική αλλαγή θα βρούμε τον τρόπο. Δεν θα λιώσω ε, σαν παγόβουνο στην Ανταρκτική, ό,τι και να πιστεύουν οι, οι αντιευρωπαϊστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Μαριάς. Στη διαδικασία Κατστία έχει το λόγο. Ο προϋπολογισμός 2020 ε, πραγματικά είναι ένας προϋπολογισμός δύσκολος και ταυτόχρονα απαιτητικός διότι γνωρίζουμε όλοι τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του brexit. πρέπει όμως να επικεντρωθούμε θα έλεγα στο πώς αυτός ο προϋπολογισμός θα ακολουθήσει πολιτικές που ενισχύουν τους νέους και τις γυναίκες. θα πρέπει να υπάρξει προτεραιότητα στην καινοτομία την έρευνα και την ανάπτυξη για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη με θέσεις εργασίας και αυτό σημαίνει στήριξη της απασχόλησης των νέων οι νέοι οι οποίοι έχουν έρθει πλέον ξανά στο προσκήνιο μια και παλεύουν για το περιβάλλον και χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις των νέων σε όλη την ευρώπη για το περιβάλλον διότι δείχνουν ένα μήνυμα αποφασιστικό οι νέοι που πρέπει να στηριχθούν με το πρόγραμμα horizon 2020 για τα ερευνητικά ιδρύματα για την ακαδημαϊκή κοινότητα για να έχουν ευκαιρίες στην εκπαίδευση για να μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότερα κονδύλια στην περίφημη πρωτοβουλία για απασχόληση των νέων και από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει όλες οι πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης να στηρίζουν τις γυναίκες και να λάβουμε υπόψη κύριε Έτιγκεν ότι θα πρέπει να ενισχύουμε τις πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης που λαμβάνουν υπόψη την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επιτέλους στην ισότητα των δύο φύλων. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για την ανοχή σας. herr präsident verehrte damen und herren abgeordnete damen und herren! κύριε πρόεδρε κυρίες και κύριοι η σημερινή σας γνωμοδότηση εμπλουτίζει την εργασία μας. Τώρα κάνουμε την προπαρασκευή εργασία για το προσχέδιο προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, το οποίο θα σας αποστείλουμε σε μερικές εβδομάδες. για να ζητήσουμε την γνώμη του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου. Και αυτά που μου λέτε με βοηθάνε για να διατυπώσουμε την πρότασή μας. Λαμβάνω λοιπόν ε, σοβαρά υπόψη τι προσδοκίε του Κοινοβουλίου λόγω των επιπτώσεων του Brexit. Και θα λάβουμε υπόψη λοιπόν τι επιπτώσει αυτέ στο προσχέδιό μας τις επόμενες μέρες. Ίσως ε, αύριο μεθαύριο να ξέρουμε περισσότερα και να είστε σίγουροι ότι το σχέδιο 2020 θα βασιστεί ε, σε τι εξελίξεις θα προκύψουν. Είτε οι φίλοι μας θέλουν να συμμετάσχουν πλήρως ε, στη διαδικασία διαμόρφωσης του προορισμού 2020 είτε αν το Brexit χωρίς συμφωνία έχει επίπτωση ότι του χρόνου δεν θα υπάρξουν πληρωμές ε, από το Λονδίνο. Αλλά και καμία συμμετοχή στα προγράμματα βέβαια. Η νομική μας άποψη δεν αλλάζει. Ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι το πλαίσιο ε, θα πρέπει να ισχύει και για τα 28 κράτη-μέλη μέχρι το τέλος του 2020. Δηλαδή αυτό που αποφασίστηκε το 2013. Πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν όλες τις νομικές δυνατότητες ούτως ώστε να γίνουν οι αναγκαίες ε, πληρωμές και να εφαρμοστούν τα δικαιώματα μέχρι το τέλος του 2020. Όμως με βάση την αρχή της πρόληψης θα πρέπει να συμποβάλουμε ένα προσχέδιο προπολογισμού το οποίο λαμβάνει επίση υπόψη την κατάσταση της Βρετανίας ε, χωρίς την συμβολή της αλλά και χωρίς τις πληρωμές πως αυτήν. Δηλαδή θα μας λείπουν 12 δις. Και αυτό το κενό πρέπει να το καλύψουμε με την πρότασή μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα μπω τώρα σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες για την εκτέλεση του προβλησμού του 2019 αλλά θα μπορούσε κάλλιστα σε λίγες ημέρες στο σώμα αυτό να φέρουμε έναν διορθωτικό προϋπολογισμό για να καλύψουμε ένα, ένα κενό 6 δισεκατομμυρίων παραδείγματος 12 ε, δις του χρόνου 6 δισεκατομμύρια φέτος και το ξέρετε όπως και εγώ το μοναδικό επίπεδο της Ευρώπης που δεν έχει δικαίωμα να δημιουργήσει χρέη είναι το ευρωπαϊκό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εκδώσουν χρέος, οι περιφέρειες το ίδιο, οι δήμοι το ίδιο. Εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την απόλυτη υποχρέωση κάθε μέρα να αντιστοιχούμε τα έσοδα με τα έξοδα. Και μας απαγορεύεται να προσφύγουμε σε δανεισμό. Θα μπορούσαμε, όπως σας είπα, επαναλαμβάνω, να ξεκινήσουμε σε λίγες μέρες διαβουλεύσεις για το πώς θα καλύψουμε 6 δισεκατομμύρια φέτος, πώς θα αντισταθμίσουμε 12 δισεκατομμύρια του χρόνου. Μόλις ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο Λονδίνο, θα έρθω να σας ενημερώσω εσάς και το Συμβούλιο. Βεβαίως, για το πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας ως Κομισιόν. Έχουμε κάνει προτάσεις για το κενό του Brexit, το οποίο θα καλυφθεί κατά 50% από περικοπές και κατά 50% από υψηλότερες εισφορές. Εάν η συνταγή αυτή σας φαίνεται λογική και δίκαιη, μπορείτε να την ακολουθήσετε και για το 2019 και 20. Δηλαδή 6 δισεκατομμύρια φέτος ενό διορθωτικού προπολογισμού θα μπορούσαν να καλυφθούν μέσω 3 δις επιπλέον εισφορών και 3 δις περικοπών. Και τα 12 δισεκατομμύρια του έτους με 6 δισεκατομμύρια περικοπές και 6 δισεκατομμύρια υψηλότερες εισφορές των κρατών. Η κυρία Νιαριάδα μου άσκησε κριτική γιατί ήμουν στο τηλέφωνο. Πράγματι, δεν μπορούσα να πιστέψω το αποτέλεσμα στη Βουλή των Κοινοτήτων, γι' αυτό έπρεπε να ρωτήσω. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι η δημοκρατία είναι αξιόπιστη όταν ε, κάνουμε κριτική, αλλά είμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε και την απάντηση. Και αντίστροφο. ο κύριος Έθριτς αφιέρωσε όλο του το αξιοσέβαστο ειδικό βάρο για να ασκήσει πολεμική κριτική για τεράστιε δαπάνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και εδώ πέρα να πω κάποια ξεκάθαρα πράγματα στους πολίτες μας. Ο κάθε πολίτης της Ευρώπης που με υδρότα ή με επενδύσεις. Βγάζει 100 ευρώ. Δίνει 50 ευρώ σε φόρους, ε, τέλη κτλ. Αυτό είναι ο μέσο όρος στην Ευρώπη. 50%. Και από τα 50 ευρώ, 1 ευρώ πηγαίνει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση. 49 παραμένουν σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη, σε Γλασκόβη, Στουτγκάρδη, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ένα από τα 50 πάει στην Ευρώπη, 49 είναι στα κράτη-μέλη, δήμους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το 1 ευρώ από τα 50 ε, θα έπρεπε να το αξίζει η Ευρώπη. Ειδικά όταν δημιουργεί προστιθέμενη αξία έτσι και η προσθέμενη αξία φαίνεται στο Erasmus υπέρ της νέας γενιάς που ε, ζει και μαθαίνει την Ευρώπη την κατάλληλη στιγμή με τα μεγάλα ερευνητικά έργα όπου απέναντι στην ε, Google και στην Silicon Valley γενικώ κανένα κράτος μέλος και κανένα πανεπιστήμιο ούτε τα καλύτερα ούτε το Cambridge και Oxford από μόνα τους δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Θα ήθελα να ελπίζω ότι οι φίλοι μας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας, όπως θέλουν οι ερευνητές σε Oxford, Cambridge και Λονδίνο, έτσι ώστε να μην καταντήσει η Μεγάλη Βρετανία, μικρή Αγγλία, στον τομέα της έρευνας. Η προσθέμενη αξία λοιπόν ο αποφασιστικός παράγων για κάθε ευρώ που επενδύουμε. Και νομίζω θα σας πείσει και η πρόταση που θα φέρουμε. Η ιδέα του βουλευτή Όλμπριχτ, πάρα πολύ σημαντική, ότι το 2020 είναι ο τελευταίος προπολογισμό του τωρινού πλαισίου και ένας προπολογισμό γέφυρα για το επόμενο πλαίσιο. Γιατί κάποια προγράμματα είναι ήδη πιλωτικά προγράμματα για το επόμενο πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας. Γι' αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας, για τον συντονισμό με την κυρία Χολμαϊρ. Οπωσδήποτε θα τα δούμε αυτά και το αργότερο την άνοιξη θα ε, δούμε τις συνέπειες του Brexit. Ελπίζω να μην είναι πολύ δραματικές, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό. Ελπίζω όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους ειδικού του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αυτού να είναι και στο επόμενο. Και για όσους δεν επιστρέψουν, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συζήτηση που είχαμε. Παραδείγματος χάρη τον κύριο Τάραντ. Θεωρώ ότι πέρα από κόμματα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρία Χολμάιερ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, πολύ καλή συζήτηση. Για το Brexit ομολογώ ότι δεν περίμενα ένα αποτέλεσμα 312 έναντι 308 με φόβησε. Γιατί το θέμα είναι αν θέλουν να προκαλέσουν χάος ή όχι. Και επειδή μιλάμε για φίλους με τους οποίους έχουμε εργαστεί και συνεργαστεί υψηρά ετών, είναι κάτι το εντυπωσιακό και θεωρώ ότι είναι ε, κάποια περιφρόνηση θα έλεγα των φίλων. Παρ' όλα αυτά αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι τελικά θα επικρατήσει η λογική γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει συμφέροντα και στην συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας ε, τελευταία ενδιαφέρεται και για πάρα πολλά είδη συνεργασίας ε, δηλαδή ξαφνικά όταν κάτι λείπει αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό ήταν. Ελπίζω λοιπόν τελικά να επικρατήσει η λογική και να υπάρχει η δυνατότητα μιας έφτακτης συνεργασίας. Να πω δύο λόγια για αυτό το οποίο είπαν οι συναδελφοί και οδησίτες. Είναι λοιπόν σημαντικό να σταθούμε απέναντι στο Συμβούλιο, να ενισχύσουμε την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό μας. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι οι πράσινοι έχουν παυλοφικά εξαρτημένα αντανακλαστικά σε κάτι τέτοια θέματα. Αλλά αυτή ακριβώς είναι λάθος πρόθεση αυτό το οποίο λέτε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες και όχι να κάνουμε δύο-τρεις φορές τα ίδια πράγματα ακριβώ να κάνουμε κοινά έργα τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε η κάθε χώρα να κάνει τις δικές της διαδικασίες διαγωνιστικές και να ξοδέψει περισσότερα λεφτά στο τέλος. Θα ήθελα επίσης αγαπητοί συνάδελφοι να έχουμε το θάρρος στα ουσιαστικά να συμφωνήσουμε και να μην ε, διαφωνούμε εντελώς. Αλλιώς δεν έχουμε πολλές θανότητες να περάσουμε κάτι απέναντι στα κρατόμελη και θα πρέπει να δούμε και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται και αυτήν ακριβώς να εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ. Με την παρέμβαση της κυρίας Χολμέιρα ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησής διάταξης σε σχέση με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η κατάσταση στην Καράγουα. Εξ ονόματος της ε, είπα της εκπρόσωπου θα παρέμβει ο Επίτροπος Μίμικα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε την κατάσταση στην Νικαράγουα και για την εξαιρετική συνεργασία τις τελευταίες εβδομάδες η Υπηρεσία εξωτερική δράση και το Ευρωκοινοβούλιο δουλεύουν χέρι με χέρι, δείχνοντα στην πράξη πώς οι διαφορετικοί θεσμοί μπορούν να δουλεύουν προς τον ίδιο σκοπό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το αξιότιμο μέλη Ραμόν Βαρέγγι για την ισχυρή δέσμευσή του και για το ότι ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Καράγουα. Η κατάσταση στην Καράγουα παραμένει... Ε, ε, σε ένταση παρά το γεγονός ότι είχε περάσει ε, το πρώτη, η πρώτη φάση της καταστολής υπάρχουν ακόμη ε, συλλήψεις, παράνομες συλλήψεις. Πολλά άτομα έχουν καταγγελίες τρομοκρατίας ότι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις. Έχουν φυλακιστεί και αυτό είναι απαράδεκτο. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι συνεχώς υφίστανται παρενοχλήσεις και ε, σε πολλούς έχει ακυρωθεί η νομική υπόστησή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφή στη καταδίκαση αυτή της κατάστασης ε, πρόσφατα στην στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων καλέσαμε τις αρχές να αποφυλακίσουν όλους τους πολιτικούς κρατωμένους και να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους και δέουσες ε, καταστάσεις έχουμε ζητήσει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να ε, εφαρμοστούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πολιτικά μέσα ε, απαντώντας στις εξελίξεις στη χώρα. Η ad hoc αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου ε, με την επικεφαλής των Ραμών Χαουρέκη ε, πήγαν στη Μανάγουα και συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση αυτών των μηνυμάτων. Χαίρομαι που κατορθώσατε να ολοκληρώσετε ένα πλήρες πρόγραμμα συναντήσεων με Οργανώσει τη κοινωνίας των πολιτών, με ανεξάρτητου δημοσιογράφους, με οικογένειε θυμάτων. Ε, επίσης επισκεφτήκατε κρατούμενου χωρί περιορισμούς και είχατε κατευθείαν ε, συζητήσει με τον πρόεδρο Ορτέγα και την σύζυγό του Ροζάουρα Μουρίγιο. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, ήταν ε, συναντήσεις πολύ συναισθηματικά φωτισμένες και χρειάστηκε πολύ κουράγιο για να οργανωθούν. Ωστόσο ήταν απαραίτητες και σημαντικές και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για τη δουλειά που έχετε κάνει. Ε, πρόσφατες εξελίξεις μας δίνουν ελπίδες και είμαι πεπισμένος ότι η δουλειά μας έχει συμβάλει στο να δημιουργήσει ένα πιο θετικό κλίμα. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση της Νακαράγουα είχε υψηλό επίπεδο συναντήσεις με τις οργανώσεις των Αμερικανικών κρατών, με κάποιους διεθνείς φορείς και την κοινότητα των επιχειρήσεων. Δεύτερον, 100 ε, ε, κρατούμενοι στάληκαν υπό κατοίκον περιορισμό. Αυτό ήταν κατόπιν αιτήματο του Ευρωκοινοβουλίου προς τον πρόεδρο Ορτέγα. Τέλος, ε, συναντήσεις με την αντιπολίτευση ξεκίνησαν στις 27 Φεβρουαρίου. Αυτές οι πρώτες συναντήσεις οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός φίλου πορείας για να ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων ε, και ο των συμμετεχόντων και των ε, διεθνών εγγυητών για να επιτευχθούν συμφωνίες. Αυτό βέβαια παραμένει ένα δύσκολο σημείο. Επίσης και οι συνθήκες σχετικά με την ε, αποφυλάκηση περαιτέρω κρατουμένων. Είμαστε διαθέσιμοι να ε, μελετήσουμε τεχνική στήριξη και διαμεσολάβηση αν αυτό καταστεί ανάγκαιο. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη, η Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως μπορεί να συμβληθούν σε αυτή τη διαδικασία ενδεχομένως. Όλες αυτές είναι ε, θετικές εξελίξεις ε, σε σύγκριση με πριν από μερικές εβδομάδες. Παραμένουμε όμως πολύ ε, προσεκτικοί. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο σοβαρά έχει λάβει υπόψη η κυβέρνηση της αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ιδιαίτερα την ελευθερία της έκφρασης και του συνέχιστε. Ε, η, παραμένει η στρατιωτική παρουσία στην Μανάγουα η αλλαγή του δικαστικού συστήματος, του φρονιστικού συστήματος και η αποφυλάκηση των 100 κρατουμένων είναι θετικό βήμα. Αλλά δεν ξεχνάμε τους πάνω από 600 κρατούμενους που παραμένουν φυλακισμένοι. Ε, σε απάνθρωπες συνθήκες συχνά και μερικοί ε, έχουν ε, κατέλθει σε απεργία πείνας. Δεν θα ξεχάσουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαδικασία και δίκαια δίκη. Γι' αυτό η αστική συμμαχία επιμένει για την αποφυλάκηση των κατμένων και τα δικαιώματά τους. Πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση ε, θα προχωρήσει για να ανταποκριθεί στα αιτήματα της αντιπολίτευσης και για να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Ε, τα ε, κόμματα στην Νικαράγουα πριν από μερικές μέρες δεν έδειξαν την βούληση να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ελπίζω ότι η ανανέωση του ανώτατου δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν θα είναι μια άλλη χαμένη ευκαιρία στην αλλαγή της πορείας. Θα πρέπει να δούμε και τη δουλειά που κάνει η αντιπολίτευση στο να μαθαίνει από τα ε, λάθη του παρελθόντος του Ιουλίου του 2013. Ελπίζουμε να ε, ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και αυτό να δώσει τη δυνατότητα στους Νικαραγανού να αντιπροσωπευθούν, να βρουν τη δικαιοσύνη και να μπορέσουν να κατέλθουν σε ελεύθερες εκλογές για την ελευθερία τη χώρα τους. Παρά τις αμφιβολίες που μπορεί να έχουμε σχετικά με αυτή τη διαδικασία, παρά ε, τις ανοιχτές και τα πολλά θύματα που ακόμη ζητούν τη δικαιοσύνη τους, θα πρέπει να ε, ενθαρρυνθούμε από τα βήματα που έχουν ήδη ληφθεί. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή ε, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και κάποια ε, ε, σημεία συγκεκριμένα έτσι ώστε να εξέλθουμε από την τρέχουσα κρίση. Οι Ευρωπαίοι εμείς επαγρυπνούμε, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και θα συνεχίσουμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε θετικά βήματα προς μια πολιτική επίλυση της κρίσης μαζί με τους διεθνείς εταίρους μας. Άρα θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την συμμετοχή σας που είναι πολύτιμη για τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κύριε Σαλαφράνκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει ένα ψήφισμα με το οποίο θα ζητήσει την αναστολή της Νικαραγούρα από τη Συμφωνία της Σύνδεσης Κεντρικής Αμερικής και ταυτόχρονα να εισηγηθούν κυρώσεις για όλους όσους ε, ευθύνονται για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. Κατά την, ε, επίστρεψη, την επίσκεψή μας τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να διαπιστώσει, όπως ε, και η ομάδα ανεξάρτητων των πυρογνώμων, ε, είπατε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην, κατάσταση στην χώρα, ότι η κατάσταση στην Νικαράγουα δεν συνάδει με τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι σημαντικό στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσής μας. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου από το Κοινοβούλιο διαπίστωνε τις δολοφονίες που είχαν υλοποιηθεί, τις συλλήψεις, τις αυθαίρετες, τα βασανιστήρια και την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ελευθερία του τύπου. Έχετε δίκιο ότι η επίσκεψη που κάναμε στις φυλακές της Νικαράγουας ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Είδαμε ε, νέους 20 ετών να έχουν καταδικαστεί σε πάνω από 30 έτη κάθριξης. Δυστυχώς, οι πληροφορίες που λάβουμε από τη Μανάγουα είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, πάνω από 600 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι γυναίκες που συναντήσαμε στη φυλακή της Εσπεράνσα ε, έχουν ξεκινήσει η απεργία πείνα λόγω κακομεταχείριση και υπήρχε κακομεταχείριση και στη φυλακή μοντέλο. Νομίζω ότι δεν θα εξυπηρετούσαμε ε, τον αγώνα μας όπως πρέπει και ότι θα προδίδαμε τις προσδοκίες του λαού της Νικαράγουας αν ανεχόμασταν την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου αυτός ο εθνικός διάλογος να ευωδώσει να ε, υπάρξει άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των πολιτικών κρατωμένων ε, να, να ε, εγγυηθούν την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την άσκηση της ελευθερίας του τύπου και να μπορέσουν να καταρτήσουν ένα οδικό χάρτη έτσι ώστε οι πολίτες της Νικαράγουας να μπορούν να πάρουν το λόγο για να καθορίζουν τη μοίρα τους. Πιστεύω, κύριε Επίτροπε, ότι σε αυτό το κοινοβούλιο έχουμε κάνει ένα έργο με πολύ μεγάλη αφοσίωση, με μεγάλη υπομονή, όμως έφτασε η ώρα, κύριε Επίτροπε, να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Δυστυχώς, η κατάσταση δεν έχει σημειώσει θετική εξέλιξη στη χώρα και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας. Αυτή την εβδομάδα στο Μικύκλιο κάναμε μία συζήτηση για έναν εφαρμοστικό μηχανισμό για την δημοκρατική ρήτρα. Είναι παραδειγματική η περίπτωση της Νικαράγουρα και παροτρύνω την Κομισιό να είναι συνεπής με την απόφαση που θα λάβουμε αύριο στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σελαφράγκα. Ο κύριος Χαουρέγγι παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Επίτροπο για τα λόγια του σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Υπηρεσία Εξωτερικής δράση στο θέμα αυτό. Θα σα εξομολογηθώ και κάτι. Είναι ότι όλη η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποσκέφθηκε για τέσσερι ημέρε στην Ικαράγουα έζησε με πολύ μεγάλη συγκίνηση τα γεγονότα και μάλιστα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια για όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Και θα ήθελα να πω ότι είμαστε μαζί με το λαό της Νικαράγουας που κλαίει τους νεκρούς του με το λαό που υποφέρει γιατί τα παιδιά του είναι στη φυλακή με το λαό που υποφέρει που υφίσταται περιορισμούς στις ελευθερίες τους. Αυτό αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση και πρέπει να καταδικαστεί. Παραβιάζεται το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Αυτό συμβαίνει στην Καράγουα και θα ήθελα να στραφώ στους συντρόφους που βρίσκονται στα αριστερά και κατέθεσαν μια τροπολογία στο ψηφισμά μας, λέγοντας να μην υπάρχουν ε, επεμβάσεις των ΗΠΑ στην Ικαράγουα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια παρέμβαση. Το πρόβλημα, κύριε Πιμέντα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι υπάρχει μια επανάσταση η οποία έχει καταστεί ολοκληρωτική το καθεστώς έχει γίνει ολοκληρωτικό. Υπήρξε μια επανάσταση που εξηγήθηκε ιστορικά και δυστυχώς ε, περιστέλει τις ελευθερίες και καταπιέζει το λαό. Εγώ πάντοτε από την αριστερά ζητούσα την ελευθερία. Ο σοσιαλισμός σημαίνει ελευθερία, πάντοτε το λέγαμε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτό το λαό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένα σοβαρό διάλογο Μακάρι να υπάρξει ένα σοβαρό διάλογο, όμω υπάρχουν τρει βασικέ συνθήκε που δεν υλοποιούνται. Η πρώτη είναι, η πρώτο όρο είναι ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Το δεύτερο όρο είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία για του επικεφαλεί των κοινωνικών κινημάτων. Και τρίτον, οι διεθνεί οργανώσει πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα. Γιατί είναι οι παρατηρητές ε, σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι αν προχωρήσει αυτό ο διάλογο θα βοηθήσει και η Ευρώπη. Και το λέω στον κομμαντάντε Ορτέγα, αν υπάρξει σοβαρός διάλογος, εμείς θα βοηθήσουμε. Αλλά αν δεν το κάνουν, αν θέλουν να χάσουν χρόνο και αν κοροϊδεύουν το λαό, τότε θα υπάρξουν κυρώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαουρέγγι. Ο κύριος Μάκερ. Eh, voorzitter, eh, commissaris. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η αντιπολίτευση στον ε, Ντανιέλ Τα έχει πολλά προσπάθεια. Ένα από αυτού είναι ο Αλέξ ε, Φαντέγκα, γνωστό αθλητή. Ω νεαρό σαντινίστα, πάλεψε στο πλευρό του Ορτέγα κατά του δικτάτορα Σομόζα, αλλά μετά άλλαξαν τα πράγματα και τώρα ο Άλεξ διαδηλώνει κατά του Ορτέγα. Τον λέγανε μαραθωνίστα, ο μαραθωνοδρόμος, τώρα τον, λένε, τον λέει τερορίστα ο Ορτέγα. Όπως εδώ πέρα και η κυρία Κόπελς, 34 ε, ετών, συμπατριώτησά μου, η οποία κρατείται στην φυλακή Λα Εσπεράνσα. Μόλις τελείωσε μια απεργία πείνας 13 ε, ημερών και βλέπετε και τα χρώματα εδώ πέρα της ε, σημαίας ε, τη γαλανόλευκη λοιπόν μου έγραψε ένα γράμμα ο Βέλγος ο πατέρας της και μου είπε να κάνω ό,τι μπορώ για να την βοηθήσω δεν είναι δυνατόν να κλείνουν το μέλλον της χώρας στις φυλακές ο Ορτέγα έχει περάσει στην άγρια καταστολή Θα πρέπει λοιπόν να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και να γίνουν δίκαιες, τίμιες εκλογές. Ο πρόεδρος Ορτέγ είπε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνει και πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στοχευμένες και ατομικές κυρώσει. Έχουμε μια συμφωνία στην οποία υπάρχουν και ρήτρε περί δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε τις αρχές μας και την υπογραφή μας. Ευχαριστώ, ο κύριος Νάρτ. Σέρχιο Ραμίλε, Χένρι Ρουί, Λουίς Καριόν, Δώρα Μαρία Τεριές, Μόνικα Βαλτοδάνο, Βίκτορ Τυράδο, Μωυσές Χασάν, Ερνέστο Καρδενάλ, Ούγο Τόρρες, Γιοκόντα Βέλη, Μπρούκλιν Ριβέρα, Κάρλος Τούνερμαν, Ουμπέρτο Ορτέγα. Όλοι αυτοί είναι ριζοσπάστες ε, αντιτιθέμενοι στην κυβέρνηση του Ντενέλ Ορτάγα. Όσοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση αυτή ε, είναι θύμα των αντιδραστικών, θα σας πω ναι, είναι οι σύντροφοί μου, οι ε, που αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας του Σομόσα και εγώ συμμετείχα στο μέτωπο. Ήταν τιμή μου να είμαι εκεί είναι ε, λοχαγοί και υπουργοί του πραγματικού ε, σαντινισμού που σήμερα προδίδεται από τον Ντανιέλ Ορτέγα. Είναι αυτή που από τη φυλακή, από τα βασανιστήρια και τις διώξεις και από τα χαρακόμματα Περασπίστηκαν την ελευθερία και τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια για την πατρίδα του στην Ικαράγουα, που είναι και δική μου.